Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε όλοι. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ πολύ να καθίσετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από δέκα ημέρες ε, η Γαλλία επλήγει με τον πλέον δύο τρόπο. Οι τρομοκράτες ε,